ψηφίσματος. Η ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών ε, έκανε τις εξής προτάσεις. Ο κύριος Ταραμπέλα θα δουλεύει στην Επιτροπή Γυναικών. Θα γίνουν μέλη των διαφόρων επιτροπών λοιπόν. Δεν υπάρχουν αντιρρήσεις. Ε, εγκρίνονται οι προτάσεις αυτές.